ότι δεν είναι και πολύ λαμπρή η παρουσία. Έχουμε μόνο τρία μέλη παρόλα αυτά. όχι, τέσσερα, τέσσερα μέλη έχουμε, όχι τρία. Ναι, ναι, και μετράω και τον εαυτό μου. Τέσσερις. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο, όσοι είμαστε εδώ, τόσο το χειρότερο για αυτούς που δεν είναι εδώ. Τι να κάνουμε. Κύριε Άνσεπ, κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Έχουμε προβλέψει να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία θέλουμε να επεξεργαστούμε. Η ψηφιακή ενιαία αγορά έχει ξεκινήσει ο τριμερούς διάλογος σήμερα στην Επιτροπή Πολιτισμού αποφασίσαμε και ψηφίσαμε για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και κάποια άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη και συζητούνται στην ε, Επιτροπή μας. Νομίζω ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι παρόμοια. Υπάρχουν δηλαδή πολλές διαφορετικές ε, απόψεις ε, για τα θέματα αυτά. Το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, το θέμα της πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το θέμα των πρωτοβουλειών από μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά, αν μπορείτε να μας κάνετε κάποια πρώτα εισαγωγικά σχόλια και ελπίζω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει να είναι ενδιαφέρουσα. Βλέπω ότι κάποιοι εντωμεταξύ φτάνουν στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έμαθα γερμανικά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και λίγο στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτά που μου λέτε στα γερμανικά. Προτιμώ παρόλα αυτά να μιλήσω αγγλικά. Δεν είναι τα οποία δεν είναι και τόσο καλύτερα από τα γερμανικά μου λέει ο Επίτροπος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για τα ζητήματα της ψηφιακής αγοράς και οικονομίας με τα μέλη της Επιτροπής σας ε, συναντιόμαστε πάρα πολύ συχνά με την κυρία Κώστα συναντήθηκαμε εχθές την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα φεστιβάλ στην Εστονία και συναντηθήκαμε και εκεί. Ένα φεστιβάλ χορού. Μιλώντας για τα ψηφιακά θέματα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πριν από δύο έτη εκινήσαμε την ψηφιακή αγορά το Μάιο καθορίσαμε μια σειρά από στόχους και υποβάλαμε 35 διαφορετικές προτάσεις συμπεριλαμβανομένων 21 νομοθετικών. Και χάρη σε επιτροπές όπως η δική σας είχαμε σημαντική επιτυχία. Η συνεργασία αυτή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τον φάκελο της ψηφιακής αγοράς ήταν εξαιρετική. Καταργήσαμε το κόστος περιαγωγής, χαμηλώσαμε το κόστος της ε, μεταφοράς των κινητών αριθμών και καθότι δεν έχουμε πλέον roaming οι πολίτες ε, που επισκέπτονται άλλες χώρες ε, θέλουν και στο εξωτερικό και όταν βρίσκονται σε διακοπές να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό τους περιεχόμενο. Το οποίο συμπεριλαμβάνει τηλεοπτικές σειρές, φιλμ, μουσική, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικές εκδηλώσεις ποδόσφαιρο που είναι πάντα πολύ σημαντικό, λέει ο Επίτροπος, όταν ταξιδεύει κανείς σε άλλη χώρα. Υπογράψαμε και την ε, συνθήκη του Μαρακές, αλλά όπως έχω ήδη ξαναπεί, τρία χρόνια αργότερα δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να την επικυρώσουμε. Έχουμε κάποιες διαθεσμικές συζητήσεις σχετικά με το ποιος έχει δικαίωμα Ποιο πρέπει να υπογράψει, τα κρατημέλη και η Επιτροπή, μόνο η Επιτροπή κτλ. Τώρα εδόθη σαφήνεια επ' αυτόν Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όμως να παράσχομαι πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε και στην πρόταση του GEOBLOCKING blocking η οποία υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα εμπορεύματα και τα αγαθά που αγοράζει κανείς online από άλλο κράτος αλλά τα κατανολώνει στο δικό του μη συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων αυτοκινήτων. Σήμερα η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επ' αυτών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση ένα 65% ολοκληρώνουν μόνο επιτυχώς τις συνδιαλλαγές τους, ένα 2% δεν καταφέρνει να έχει πρόσβαση λόγω λανθασμένων ε, διευθύνσεων IP πολίτες από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία ή από οποιοδήποτε άλλη χώρα, το 25% δεν μπορεί, καταφέρνει να καταχωριστεί. Διότι και πάλι υπάρχει κάποιο λάθος ηλεκτρονικής διεύθυνσης, IP, το 30% αντιμετωπίζει προβλήματα παράδοσης με τη διεύθυνση αλλά και το 26% από τους πολίτες που επιθυμούν να αγοράσουν online από άλλη χώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το αντίτιμο διότι λαμβάνουν ένα μήνυμα ότι η πιστοτική τους κάρτα για παράδειγμα έχει εκδοθεί σε λάθος χώρα. Δεν είναι αυτή η ενιαία ψηφιακή αγορά εν ολίγης που θα επιθυμούσαμε να έχουμε. Έχουμε και τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων Η Επιτροπή Τζούρι βλέπω με έκπληξη ότι ηγείται στο φάκελο αυτό ενώ το θέμα είναι καθαρά θέμα πολιτισμού και διαφορετικότητες. Αλλά θα χρειαστούμε την δική σας φωνή και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ακουστεί η δική σας φωνή αλλά σχετικά με την οδηγία για τα πνευματικό, πνευματικά δικαιώματα, με πρέπει να συζητήσουμε, να λάβουμε υπόψη μας και αυτό το value cap. Έχουμε διαφορετικές πλατφόρμες επί τη βάση της καταχώρησης, 40 εκατομμύρια εγγεγραμμένους το μήνα και καταβάλουν σημαντικότατα ποσά στους δημιουργούς, παράδειγμα στους μουσικούς. Υπάρχουν όμως και πρόσθετα έσοδα από τις διαφημίσεις με ένα δισεκατομμύριο επισκέψεις το μήνα. Αλλά συνεισφέρουν μόνο 640 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Επομένως από, από τα 2 δις φτάνουμε στο 0,6 και η μουσική, μεταξύ άλλων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους διότι δεν λαμβάνουν επαρκείς αποζημιώσεις. Χάνουμε λοιπόν όγκο περιεχομένου τη στιγμή και την οποία δεν μπορούμε τους δημιουργούς να τους αποζημιώσουμε καταλήλως. Έχουμε και τα δικαιώματα δημοσίευσης όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες απόπειρες στην Ισπανία και στη Γερμανία ίσως όχι τόσο επιτυχείς απόπειρες αλλά οι εκδότες θεωρούν ότι εάν υπήρχε ένας ενιαίος κανόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα βοηθούσε στο πεδίο των εκδόσεων των δημοσίευσεων Επίσης, είναι μια σημαντική δήλωση και δέσμευση της Επιτροπής είναι ότι τα hyperlink θα παραμείνουν ως δικαίωμα. Και δεν μιλάω για ένα hyperlink προς φορολόγηση ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα ζήτημα επί του έχουμε και πλήρη και αξιόλογη νομολογία. και τα hyperlink ήδη καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά οι εκδότες, οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι, όλοι αυτοί ενέχονται στο θέμα αυτό. Όταν όμως τη δεκαετία του 60 οι δισκογραφικές εταιρείες έλαβαν τα δικαιώματα neighboring τα συγγενικά εν περιπτώσει δικαιώματα ήταν ένα προηγούμενο το οποίο όμως δεν τηρήθηκε για τις σημερινές ψηφιακές πλατφόρμες. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι κάποιος χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της πνευματικής του ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση. Αυτά λοιπόν τα neighboring rights θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα πιο ισότιμο παιχνίδι, ένα ισότιμο πλαίσιο κανόνων. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε και σε σχέση με το θέμα των συγγενικών αυτών δικαιωμάτων. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι αμφίσιμη η πρόταση. Το data mining, επίσης σημαντικό θέμα. Πρέπει να παράσχουμε στους ερευνητές και τους επιστήμονές μας αυτό το σημαντικό εργαλείο. Υπάρχουν τακτικές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων επί τη βάση τέξτ κειμένου, δηλαδή υποκλοπής κειμένου και δεδομένων. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο από τους πιο φιλελεύθερους κανόνες που υπάρχουν επί του θέματος αυτού. Κάποιοι ζητήν ακόμα πιο φιλελεύθερες ή ελεύθερες ρυθμιστικές διευθετήσεις από αυτές που χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο Όμως γιατί να καταστρέψει κανείς ένα επιχειρηματικό πρότυπο το οποίο λειτουργεί σωστά. Μιλούμε για σχέσεις μεταξύ των εκδόσεων των φαρμακευτικών εταιριών μεταξύ άλλων κτλ. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τους κατόχους των δικαιωμάτων, τους δημιουργούς. Η δική μας πρόταση για το text και data mining είναι ακόμα πιο φιλελεύθερη από τους κανόνες τους Βρετανικούς. Αλλά δεν θα ήταν λογικό να δημιουργήσει κανείς ένα χάος, μια αβέβαιη κατάσταση, λέει ο Επίτροπος. Ο διευθυντής σας των οπτικοακουστικών θεμάτων και η κυρία Κάμερβερτ είναι υπεύθυνη για το φάκελο αυτό και τον παρακολουθούν. Και ελπίζω με τους πέντε τριμερείς διαλόγους που θα έχουμε να βρούμε και επ' αυτού συνένεση. Είμαι σχεδόν ικανοποιημένος με τη διαδικασία, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά στα κράτη-μέλη, γιατί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχουν προκύψει κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που δηλώνουν μη ικανοποιημένες Εμείς προσπαθήσαμε να οικοδομήσουμε μια συνένεση και μια κοινή προσέγγιση. Αν κάποιος δηλώνει απογοητευμένος, τότε αυτό μάλλον δεν είναι καλό σημάδι, λέει ο Επίτροπος. Πρέπει να μιλήσουμε και για, τον, για το πρόγραμμα των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης που είναι σημαντικό θέμα και για την Επιτροπή σας, η πρωτοβουλία Creative Europe είναι σημαντική. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι θα γίνει με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Λόγω του Brexit έχουμε κάποια αβεβαιότητα, λέει ο Επίτροπος. Και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το επίπεδο του επομένου που-δου-πού. αλλά Σίγουρα πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στα μέσα επικοινωνίας. Στην Digital Europe από 100 εκατομμύρια το έτος πηγαίνουν σε προγράμματα μέσων επικοινωνίας και αυτά είναι πραγματική στήριξη στην κινηματογραφική μας βιομηχανία και χάρη στους πόρους αυτούς μπορούν να ανταγωνίζονται άλλα κέντρα παραγωγής κινηματογραφικής στον κόσμο. Επίσης έχουμε το θεματοφυλάκιο των ψηφιακών δεξιοτήτων επί τη βάση του οποίου τα κράτη-μέλη πρέπει, και η πλειοψηφία της το έχει κάνει, να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές επ' αυτού. Με την πρωτοβουλία λοιπόν αυτή υπάρχει μια κοινή κατανόηση σχετικά με το ότι οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι κάτι το εκπληκτικό και άγνωστο, είναι βασικές και απαιτούμενες δεξιότητες. Με την επόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής μας, της στρατηγικής μας, εντοπίζουμε και νέες περιοχές εστίασης και εδώ μιλώ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για την οικονομία των δεδομένων και για τις πλατφόρμες. Θέμα το οποίο βεβαίως σχετίζεται με την Επιτροπή σας. Σήμερα μιλούμε για τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των πλατφορμών. Οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις είναι δυσαρεστημένες διότι λένε ότι δεν έχουν ισότιμους κανόνες διαπραγμάτευσης με τις μεγάλες κλίμακας ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και τους είναι δύσκολο να καταλάβουν επί τη βάση ποιών κανόνων αφαιρούν από τους καταλόγους τους συγκεκριμένες μικρές επιχειρήσεις. και επομένω πώς να προωθήσουν τις δικές τους υπηρεσίες. Πώς να βρει κανεί αυτά τα αποτελέσματα αναζήτησης ώστε να αναδυθούν άλλες επιχειρήσεις στην αγορά. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις πρακτικές στην οικονομία και επίσης όταν μιλούμε για μηνύματα μίσους ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτήν την αρχή βάσει της οποίας και η οδηγία, η οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου δεν επιτρέπει την παρακολούθηση του ψηφιακού περιεχομένου, αλλά υπάρχει μια ειδοποίηση, υπάρχει μια υποχρέωση ειδοποίηση. Το τι βέβαια σημαίνει αυτή η αρχή, duty and care principle σημαίνει απλώς ότι τσεκάρουμε ένα συγκεκριμένο πεδίο με διεύθυνση κατοικία ή ηλεκτρονική είναι ασαφές. Και ποιος θα αντιδράσει για να πει ότι ναι, λάβαμε την ειδοποίησή σας εντός ποιου χρονικού διαστήματος πρέπει οποιοδήποτε αρμόδιος φορέας να πει «Μάλιστα, το γνωρίζουμε, το παρακολουθούμε» ή «Είναι νόμιμο, δεν παραβιάζει τους κανόνες, θα παραμείνει». Ή αν έχω αναφορτώσει κάτι σε μια πλατφόρμα που κατά την ενημέρωσή μου ήταν 100% νόμιμο, ενώ κάποιος άλλος εναλαμβάνει δράση για να αφαιρέσει το περιεχόμενό μου από την πλατφόρμα. Εγώ τι δικαιώματα έχω για να προστατεύσω τα συμφέροντά μου. Είναι ασαφές και θέλουμε να φέρουμε σαφήνεια σε αυτά τα θέματα. Μιλώντας για την οικονομία των δεδομένων πρέπει να μιλούμε για την ελεύθερη ροή τους. Σήμερα η κατάσταση στην Ένωση Έχουμε 56 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, λέει ο μιλητή, το οποίο σημαίνει ότι είναι απλά ένα αδιέξοδο. Είναι πιο εύκολο να συλλέγονται τα δεδομένα και να παραμένουν εντός της αυτής χώρας, αλλά έτσι παρεμποδίζουμε την καινοτομία, παρεμποδίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις. οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν 28 κέντρα εδωμένων σε 28 χώρες, αλλά για τις νέες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις είναι απολύτως αδύνατον. Και το μήνυμα προς τα startups, προς τις νέες και μικρές επιχειρήσεις θα είναι σαφές. Μην κάνετε τίποτα ή πάτε στις Ηνωμένε Πολιτείες που έχει ελεύθερη οικονομία και προοδευτικούς κανόνες. Αν καταφέραμε λοιπόν να άρωμε τα εμπόδια της ελεύθερης ροής δεδομένων, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σημαντική επένδυση ακόμα και το ύψος των 4 δις, η οποία όμως θα επιφέρει 8 δις μέσω της καινούργιας οικονομίας. Τώρα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που έχει σχέση με όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου και όχι μόνο με τη δική σας, η συνεργασία μεταξύ των εγκληματικών οργανωμένων ομάδων είναι μια πραγματικότητα. Η συνεργασία όμως μεταξύ των νομικών διοικήσεων, διοκτικών και άλλων δεν είναι τόσο σαφής και επομένως δεν έχουμε ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ αυτών. Και οι κακοί πάντα είναι σε θέση να έχουν και καλύτερη νομική υπεράσπιση από τους καλούς. Γι' αυτό κινήσαμε μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από το 2013 Οπότε κάποιο θα μπορούσε να πει τέσσερα χρόνια λοιπόν και τώρα ήδη σκέπτεστε τη νέα στρατηγική. Ναι, αλλά η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Το 2013 καλά-καλά δεν είχαμε το διαδίκτυο των πραγμάτων Όμως μέσω των διασυνδεδεμένων συσκευών και προγραμμάτων μπόρεσε να γίνει επίθεση ακόμα και στους μεγαλύτερες κλίμακας παρόχους στον κόσμο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα πολύ αυτά σοβαρά θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, Προεδρέ, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις στις οποίες θα απαντώ απλά ναι ή όχι, λέει ο Επίτροπος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. του όντω το ρολόι μου, γιατί έχουμε διαρθρωμένο διάλογο, ξέρετε, που σημαίνει βασικά ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των Ευρωβουλευτών. Και μα είπατε κι εσεί άλλωστε ότι πρέπει να αποχωρήσετε στι 4 και 20. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλω να διασφαλίσω ότι όντω θα λάβει χώρα και ένα διάλογο μετά την παρουσίασή σα. Να δώσω τώρα πρώτα το λόγο στους συντονιστές μας για 2 με 3 λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια το λόγο μπορούν να πάρουν τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπής. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα για το διαρθρωμένο αυτό διάλογο. Χαίρομαι πραγματικά πολύ που άκουσα όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, γιατί όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς επίσης και όσον αφορά άλλα ζητήματα. Και βεβαίως όταν πρόκειται για θέματα περιεχομένου, εδώ άσχετα από την αξιολόγηση που μπορούμε να κάνουμε από γεωγραφικής απόψεως, όταν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για θέματα δημιουργών, περιεχομένου, θα πρέπει πραγματικά να δούμε όλες αυτές τις ε, συγκεκριμένες προδιαγραφές που αφορούν ε, τον γεωαποκλεισμό, τις ε, διάφορες ε, δυνατότητες να υπάρξει μια ρήτρα αναθεώρησης. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της προστασίας του περιεχομένου με όλες τις ε, διασφαλίσεις βέβαια που θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι ώστε η πολιτισμική πολυμορφία και για τις κινηματογραφικές ταινίες αλλά και για τους άλλους τομείς να αρχίσει πραγματικά να ισχύει και να αναπτύσσεται. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Δεν έχω ακούσει για το θέμα αυτό της ε, εδαφικότητας κάποια συγκεκριμένη θέση από την Επιτροπή. Κυρία Κώστα. Σε ευχαριστώ Πέτρα και συγχαρητήρια γιατί σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τους εκπροσώπους Εστονικής Προεδρίας και είδα και τον Επίτροπο Άνσιπ στο Τάλιν και είχαμε ήδη κάποια πρώτα πολύ θετικά δείγματα. Τώρα όσον αφορά τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, πολύ θετικά τα πρώτα δείγματα, εκπροσωπώντας όμως την Επιτροπή Πολιτισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε μια ισορροπία όσον αφορά την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των πολιτών στο νέο αυτοψηφιακό περιβάλλον. Πριν από λίγο και εκπρόσωπος του ΕΛΚ είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική πολυμορφία. Ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει, να αναγνωρίσουμε όχι μόνο τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, αλλά να έχουμε και την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή του πολιτισμικού περιεχομένου και την προστασία και την πρόσβαση σε αυτό στη συνέχεια. Όλα αυτά τα οποία είπατε, η δυνατότητα μεταφορά του περιεχομένου αυτού, ανάγνωσή του από τη μία χώρα στην άλλη, η κατάργηση των τελών περιαγωγή, όλα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Δύο σημαντικά ζητήματα όμω τώρα. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώ επίση και ο νέο αυτό κώδικα, ε, η νέα αυτή συμφωνία στην οποία αναφερθήκατε, όσον αφορά την ειδοποίηση, το σύστημα αυτό ειδοποίησης, ήδη από το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να το έχουμε, θα αρκεστούμε απλώς σε μια συμφωνία διοργανική ή θα πάρει μια πιο επίσημη μορφή μέσω κανονισμού, μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Θα έχουμε έναν κώδικα δεντολογίας όσον αφορά τον ψηφιακό κόσμο. Έπειτα, όσον αφορά την προστασία στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να καταφέρουμε να προστατεύσουμε και τους ανήλικους, τα παιδιά. Πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή αν έχουμε όντως αξιολογήσει τους μεγαλύτερους κινδύνους που εμφανίζονται στο ψηφιακό περιβάλλον και να ασχοληθούμε όχι μόνο με το πολιτισμικό περιεχόμενο αλλά και με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επίσης, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Κάναμε πολλές συζητήσεις για το ζήτημα αυτό όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικών περιεχομένων. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε ότι η πολιτισμική παραγωγή, η κινηματογραφική για παράδειγμα παραγωγή, πολλές φορές περιορίζεται στη γεωγραφική επικράτεια συγκεκριμένων κρατών μελών, ενώ είναι δύσκολη η πρόσβαση από άλλες χώρες ή η εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος σε κάποιες άλλες χώρες. Προβλέπετε εσείς κάποια άλλα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγής ώστε να καταφέρουμε τελικά να έχουμε μια καλύτερη μεταφορά των έργων αυτών από τη μία χώρα στην άλλη προστατεύοντας παράλληλα τα πνευματικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Για να το... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο της Εστονίας. Είχαμε δύο υπουργούς από την Εστονία το πρωί, τώρα έχουμε έναν επίτροπο από την Εστονία. Θα ήθελα παρόλα αυτά να θέσω ένα ερώτημα, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσίασή σας, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τα πνευματικά δικαιώματα. Στο παρελθόν ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοστικών μέσων και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με διαφορετικούς τρόπους να εισάγουμε διατάξεις όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα. Είχαμε το γεωγραφικό αποκλεισμό, είχαμε πολλά άλλα στοιχεία τα οποία φτάνουν σε εμά από άλλες διαφορετικές επιτροπές. Πολλές φορές υπάρχει και μια επικάλυψη, για παράδειγμα, ο ορισμός όσον αφορά τις πλατφόρμες ανταλλαγής ε, οπτικοκουστικού περιεχομένου, video sharing platforms, ή όσον αφορά το περιεχόμενο το οποίο παράγουν οι χρήστες, πώς ακριβώς ορίζεται αυτό. Πολλές φορές ορίζεται με εντελώ διαφορετικό τρόπο όταν μιλάμε για τις πλατφόρμες αυτές και με εντελώ διαφορετικό τρόπο όταν μιλάμε για την ε, οδηγία ε, οπτικοκουστικών μέσων. Ουσιαστικά έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες ξεκινούν από πολλές διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και καταλήγουμε τελικά σε μια πλήρη σύγχυση. Εδώ πέρα τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά όλες αυτές τις πτυχές που έχουν να κάνουν τελικά με το χώρο του διαδικτύου. Εσείς έχετε εντοπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και θεωρείτε ότι μπορούμε τελικά να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο προκειμένου να έχουμε και μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ. Κύριε Άντσιπ, σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε όλες αυτές τις προτάσεις. Θα ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Την τελευταία δεκαετία έχουμε τα ίδια και τα ίδια και συζητάμε εδώ ελευθερία στο διαδίκτυο, όλες αυτές οι ελευθερίες και βεβαίως να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος να ρυθμίσουμε τις δυνατότητες αυτές και τις πλατφόρμες. Στα γερμανικά μιλάμε για μια έξυπνη ρύθμιση. Υπάρχουν διαφορετικά σημεία από τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και γι' αυτό και θα αναφερθώ σε τρία σημεία τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Είπατε ότι θέλουμε να υπάρχει, και αυτή είναι η θέση της Επιτροπής, ελεύθερη σύνδεση, free linking. Το θέμα τώρα των πνευματικών δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο τους Ευρωπαίους δημιουργούς. Υπάρχει και η δίκαιη κατανομή αυτών των πλέον εκτιμάτων και κυρίως θα πρέπει να σκεφτούμε και τους δημοσιογράφους. Το θέμα τώρα της εδαφικότητας, το θέμα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο θα είναι το μοντέλο το οποίο θα επιλέξουμε για την χρηματοδότηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστρέψουμε το υπάρχον σύστημα χρηματοδότησης Αναφερθήκατε στον ε, γεωποκλεισμό και στον μη δικαιολογημένο γεωαποκλεισμό. Υπάρχει όμως και δικαιολογημένος και μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράμετροι που θα επιλέγατε. Τώρα, το θέμα του value gap. Από την άποψή μου πρόκειται για κάτι που αφορά κυρίως τις τρευλώσεις στον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Το θέμα των ε, μεγάλων αμερικάνικων ε, επιχειρήσεων, Google ε, και άλλων, που έχουν παρουσία στην Ευρώπη χωρίς να συνεισφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν βεβαίως πολύ συγκεκριμένοι ε, λόγοι για τους οποίους εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιλέγετε μία πιο επιθετική στάση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλο να θέλει να κάνει ερώτηση. Θα σας κάνω εγώ μια πολύ σύντομη ερώτηση. Λοιπόν, μιλήσατε για τις δεξιότητες ε, της ψηφιακής ε, αγοράς, ψηφιακές δεξιότητες τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετή, ε, νομοθετικού περιεχομένου ή όχι για το θέμα αυτό. Α, δεν σας είδα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα. Μόνο και μόνο για να σας εκθέσω την άποψη που έχουν πάρα πολύ πλέον από αυτά τα οποία διαβάζουμε στις εφημερίδες, αλλά για να εκφράσω και μια προσωπική άποψη, η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Πώς είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούμε την καταπληκτική αυτή ευκαιρία που μας δίνουν οι ψηφιακές πλατφόρμες πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των πλατφορμών αυτών, όχι μόνο όσον αφορά τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, αλλά και όσον αφορά τις α, πληροφορίες εκείνες οι οποίες είναι εντελώ τέλεια κατασκευασμένες, οι οποίες όμως στη συνέχεια συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση, στον αποπροσανατολισμό και τελικά συμβάλλουν σε μία πληροφόρηση η οποία είναι εντελώς, εντελώς παραπλανητική. Εγώ είμαι παιδίατρος, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της υγείας και θα ήθελα να σας ρωτήσω το ακόλουθο. Πώς μπορούμε παράλληλα με την απόλυτη ελευθερία στο διαδίκτυο να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να μας προστατεύει από την διάδοση ειδήσεων που θα μπορούσαν τελικά να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνε όσον αφορά κάποια ευάλωτα άτομα. Οι νέοι, για παράδειγμα, οι οποίοι ενδεχομένω να διαβάζουν σε σχέση με οικονομικά ζητήματα πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Ο Λουίτζο Μοργάνο έχει το λόγο. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εγώ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω πολύ σύντομα, κύριε Πίτροπε. Πρώτον, όσον αφορά την ψηφιακή αριστεία, ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους. Το πρόβλημα έγκυται κυρίως στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Επομένως, ποιες είναι οι δράσεις που θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτό. Δεύτερον ερώτημα από το Μάρτιο του 2017 το Ευρωπαρόμετρο έκανε μία έρευνα όσον αφορά τις επιπτώσεις της ε, ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τα αποτελέσματα τι καταδεικνύουν, ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή βλέπουν ε, θετικά την επίπτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία, την οικονομία, την ποιότητα της ζωής, ε, και εν γέννη δείχνουν εμπιστοσύνη στις νέες ευκαιρίες που μας επιφυλάσσουν οι νέες αυτές τεχνολογίες. Διαφαίνονται όμως και δύο επικριτικές στάσεις σε αυτή τη μελέτη, σε αυτή την έρευνα. Οι συμμετέχοντες καταρχάς είπαν ότι είναι απεσιόδοξοι σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης. 7 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η ρομποτική, τα ρομπότα, το artificial intelligence πρόκειται και ουσιαστικά να οδηγήσει σε μείωση των θέσεων απασχόλησης για τους ανθρώπους. Και σε σχέση με αυτό διαφαίνεται και άλλη μια άποψη. Σε σχέση με το 2014 είναι λιγότεροι οι Ευρωπαίοι αυτοί πολίτε, οι οποίοι θα θέλανε να έχουν στο χώρο εργασία του ένα ρομπότ ή τουλάχιστον κάποιε αρμοδιότητε να ληφθούν από τα ρομπότ. Και τίθεται ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα τη εμπιστευτικότητα, του απορρίτου, τη ιδιωτική ζωή. Ασφάλεια και ιδιωτική ζωή είναι δύο ζητήματα τα οποία είναι ανηλένδετα και θα ήθελα για αυτά να μας δώσετε δυνατόν κάποιες περισσότερες πληροφορίες πάντα σε σχέση με τις θεματικές αυτές ενότητες τις οποίες θα επεξεργαστεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τζούλη Γόρτη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δύο σημεία θα ήθελα να δείξω. Γυναίκες και οι νέοι. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρετε έτσι ώστε να ενισχύσετε την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο. Ξέρουμε ότι, ότι έχει σχέση με μαθηματικά, με επιστήμες, με μηχανικές ε, επιστήμες. Οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται αρκετά. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Δεύτερον, οι νέοι Κατά κάποιο τρόπο ο ψηφιακός κόσμος ανήκει στους νέους, ε, δεν το φοβούνται, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτόν και ε, είναι αυτοί που πραγματικά εποφελούνται από την καινοτομία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τους ακούμε, είμαστε ανοιχτοί σε αυτούς και τι ευκαιρίες τους δίνουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν περισσότερο και να τους προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες ε, στον κόσμο το ψηφιακό και όσον αφορά την αγορά εργασίας. Εγώ συνεργάζομαι με ομάδες νέων από πέρσι και πραγματικά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες στον ψηφιακό κόσμο για τους νέους. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πάρα πολλές ερωτήσεις και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, έτσι δεν είναι. πώ θα καταφέρουμε να βρούμε χρόνο όμω για δεύτερο γύρο συζήτηση, αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, Α ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση, IGF και Nay. Το ζήτημα αυτό ετέθηκε εχθές και σα είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας να διοργανώσουμε μία συνάντηση με τους ανθρώπους της IGF και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδάξουμε τις ψηφιακές δεξιότητες ήδη από τον υπηαγωγείο. Μαθήματα coding θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των σχολικών προγραμμάτων σε όλα τα σχολικά επίπεδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αναφερθήκατε σε συγκεκριμένε δράσει που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να στοχεύσουμε κυρίω του ε, νέου. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή την Code Week, ε, μια εβδομάδα coding στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων νέων. Δεκάδες χιλιάδες έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτές τις εβδομάδες coding. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερους νέους. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει το στερεότυπο ότι είναι μόνο κάποια gigs που ασχολούνται μόνο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ασχολούνται με το coding. Ανταυτού νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο την εικόνα πολλών αγοριών και κοριτσιών που ανεξάρτητα από τις γνώσεις που έχουν στις ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι πλέον σε θέση να δημιουργούν τα ίδια βιντεοπαιχνίδια και είναι μόνο 8, 9 ετών, 12 ετών. Πρόκειται για πολύ νέα παιδιά ουσιαστικά και αυτά ακριβώς θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να αποκτήσουν τις ψηφιακές αυτές δεξιότητες το συντομότερο δυνατό, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Πολύ συχνά όμως θεωρούμε ότι οι πιο μεγάλοι, οι πιο ηλικιωμένοι βρίσκονται πια σε μια πολύ προχωρημένη ηλικία και δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτή η στάση είναι εντελώς λαθασμένη. Και οι μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι πολίτε είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν όλε αυτέ τι καινοτόμε λύσει που προσφέρει το διαδίκτυο, αρκεί βέβαια οι λύσει αυτέ να είναι φιλικέ προ το χρήστη. Αν το εξασφαλίσουμε αυτό, τότε όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο και όλο και περισσότεροι πολίτες θα αποζητούν τις ίδιες ψηφιακές λύσεις και από άλλα όργανα και από άλλους παρόχους υπηρεσιών τώρα. Ισότητα των δύο φύλων ιδίως όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής. Θα έλεγα ότι ένα 80% των ανθρώπων που εμπλέκονται στον τομέα της πληροφορικής είναι κυρίως άνδρες. Ενώ ένα 20% μόνο είναι γυναίκες. Οι γυναίκες εργαζόμενοι όσον αφορά συγκεκριμένα τον κλάδο, τον επαγγελματικό κλάδο της πληροφορικής. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες προκειμένου να μπορούν να εξορροπούν καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερα το επαγγελματικό περιβάλλον προκειμένου να θαρρύνουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να εργάζονται στο μέσο της πληροφορικής. Αυτό ισχύει και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ συχνά υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι πολύ διστακτικοί ή ακόμα και φοβούνται μπροστά στην επέλαση της νέας ψηφιακής εποχής, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Και υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη εν γέννη θα μας αρπάξουν τις δουλειές μας, θα χάσουμε τις θέσεις απασχόλησής μας και το καθεξής. Εγώ πιστεύω πραγματικά στην πρόοδο. Η πρόοδος ανέκαθεν δημιουργούσε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πριν από 100 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 1,5 εκατομμύρια γεωργούς. Σήμερα έχουν μόνο 800.000 περίπου γεωργούς, αλλά από άποψη παραγωγής αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η παραγωγή αυξήθηκε πάρα πολύ γρήγορα τα τελευταία αυτά χρόνια και η αποδοτικότητα αυξήθηκε ακόμα πιο γρήγορα στις ΗΠΑ. Πριν από 10 χρόνια στις ΗΠΑ είχαν 699.000 ανθρώπους που εργάζονταν με μηχανές φάξ, Πόσα, πόσους ανθρώπους έχουν αυτή τη στιγμή που εργάζονται με μηχανές φάξ. Πολύ λιγότερους προφανώς. Εγώ πιστεύω λοιπόν στην πρόοδο και να σας δώσω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Κάθε φορά που αγόραζα μια καινούργια ηλεκτρονική συσκευή, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ, ένα iPad κτλ. Πάντα μπορούσα και εργαζόμουν περισσότερο. Γινόμουν όλο και πιο διαθέσιμος. Και το ίδιο νομίζω ισχύει και για εσά. Οι νέε τεχνολογίε μα δίνουν τη δυνατότητα να εργαζόμαστε περισσότερο και να είμαστε πιο διαθέσιμοι. Επομένω, σα μην θεωρούμε ότι θα χάσουμε τη δουλειά μα και ότι θα έρθουν τα ρομπότ να μα αρπάξουν τι θέσει απασχόλησή μα. Όσοι παρόλα αυτά ανησυχούν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους εν μέρη, οι φόβοι τους μπορεί να είναι κάπως βάσιμοι και σίγουρα ορισμένοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Τα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι εθνικές αρχές, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, τα εργοστάσια, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αποδεχθούν αυτή την ε, διαδικασία διαβίου μάθησης σε μια αναπόφευκτη πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή αποτελεί απλώς ένα σλόγγαν, αλλά πρέπει να γίνει μια απτή πραγματικότητα, διότι σε ορισμένους τομείς σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά τους. Και πολύ συχνά Ορισμένοι προβάλλουν και κάποιες ιδέες ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας φόρος για τη χρήση ρομπότη, φόρος για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ε, μα δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Όσον αφορά για παράδειγμα κάποια μαθήματα τα οποία παρακολουθώ εγώ. Έχω ένα δάσκαλο και μία δασκάλα, προσπαθούν να μου διδάξουν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας. Νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιοι όροι σας διαφεύγουν ή κάποιες δεξιότητες σας διαφεύγουν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρησιμοποιώ εγώ στο iPad μου, γιατί όπως καταλάβατε ο δάσκαλος αυτός και η δασκάλη είναι καθαρά εικονική. Κάθε φορά λοιπόν που Προσπαθώ εγώ να κάνω επανάληψη στα γαλλικά μου. Κάθε φορά που ξεχνάω μια γλώσσα, συγγνώμη, έναν όρο, μια λέξη, εμφανίζεται αυτός ο δάσκαλος και δασκάλα και μου λένε η λέξη η οποία θυμάσαι είναι η κτλ. Πώς μπορούμε να φορολογήσουμε αυτούς τους εικονικούς βοηθούς, πώς μπορούμε ουσιαστικά να φορολογήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το φορολογήσουμε, αλλά είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Νομίζω λοιπόν ότι κάθε φορά που ακούγονται ιδέες αυτές για τη φορολόγηση των ρομπότ, ουσιαστικά αν το κάνουμε αυτό θα δημιουργήσουμε εμπόδια σε όλες αυτές τις ε, καινοτόμες διαδικασίες. Και ας μην ξεχνάμε, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία αυτή και μάλιστα έχει αναπτύξει και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Απομένει σε εμά να δούμε αν θα μπούμε πάνω στο τρένο αυτό το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, θα μείνουμε εκτό. Μιλάμε για παγκόσμιε συνθήκε ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε εμεί να σταματήσουμε και να μαχαιτήσουμε την πρόοδο. Αν λοιπόν εμεί δεν χρησιμοποιήσουμε τα ρομπότ, κάποιο άλλο θα το κάνει για μα κάπου αλλού. Τα ρομπότ αυτά υπάρχουν ούτως ή άλλως. Στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ήδη χρησιμοποιούνται ρομπότ και μάλιστα ο αριθμός κατά κεφαλήν είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη ξέρουμε ότι μόλις χρησιμοποιούνται τόσο πολλά ρομπότ στη Γερμανία, το ποσοστό ανεργίας είναι από τα πιο χαμηλά στη Γερμανία. Χάρη στα ρομπότ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι Μπορούμε να προωθήσουμε κάποιες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η υπεργολαβία για παράδειγμα, η μετάθεση κάποιων εσωτερικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικές εταιρείες ήταν κάτι το οποίο πάρα πολύ πριν από κάποια χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ρομποτική μπορεί να αναλάβει ένα τμήμα των υπηρεσιών που στο παρελθόν ανήκαν στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Και Στη Γερμανία, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι η δημιούργησε ένα νέο εργοστάσιο και δεν απέλησαν κανέναν. Αλλά στα πλαίσια της παραγωγής χρησιμοποιούν και ρομπότ και αυξήθηκε πάρα πολύ παραγωγή και χάρη στα ρομπότ. Να λοιπόν ένα πολύ θετικό παράδειγμα ανάθεσης κάποιων αρμοδιοτήτων σε ρομπότ. Ας μην φοβόμαστε λοιπόν τη ρομποτική, Εμεί μην φοβόμαστε την ψηφιοποίηση, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο είναι οι ίδιοι οι πολίτες και οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και όχι μόνο οι νέοι. Τώρα όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσει. Προφανώς το ζήτημα είναι επίκαιρο, καυτό, παντού, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ιδίω οι πλατφόρμες αυτές ε, τις οποίες αναφέρατε, αυτές θα πρέπει να σας απασχολήσουν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές, τις πλατφόρμες που διαδίδουν ε, ψευδείς ειδήσει, αλλά και εμείς εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό των πλατφορμών. Αν οι πολίτες δεν εμπιστεύονται αυτές τις πλατφόρμες, ε, δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Έτσι δεν είναι. Πριν από δέκα χρόνια, στη χώρα μου, στην Εστονία, υπήρχαν ορισμένες εφημερίδες που το 90% βασικά του περιεχομένου τους το βάζανε σε ιστοσελίδες και τα περισσότερα βέβαια άρθρα συνοδεύονταν από ανώνυμα σχόλια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό βασικά των σχολείων ήταν ανυπόγραφα. Καταλαβαίνετε όμως ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν ποτέ να εμπιστευθούν όλα αυτά τα άρθρα, όλα αυτά τα σχόλια τα οποία ήταν ανυπόγραφα ουσιαστικά και ανώνυμα. Βλέπαμε λοιπόν ότι στο παρελθόν οι εφημερίδες αυτές οι οποίες λειτουργούσαν μόνο στο διαδίκτυο και είχαν ε, ανώνυμα τελικά άρθρα, είχαν 90% ε, άρθρων, 10% παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω δεν έχουν καν τα σχόλια αυτά. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαβάζει καν τις εφημερίδες αυτές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι αναξιόπιστες αυτές εφημερίδες ουσιαστικά με την πάρδο του χρόνου χάσαν τελικά και τον αγνωστικό του κοινό. Αργά ή γρήγορα λοιπόν οι πλατφόρμες αυτέ θα πρέπει να ασχοληθούν και με το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων. Αργά ή γρήγορα πιστεύω όμω ότι θα χάσουν ούτω ή άλλω τον αγνωστικό του κοινό γιατί οι πολίτε θα σταματήσουν να τι εμπιστεύονται και εμεί όμω ω πολιτικοί θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Γι' αυτό το λόγο θα υποβάλουμε μια πρόταση όσον αφορά την αρχή του duty of care, το ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτή η δέουσα επιμέλεια και να υπάρχει και ένα σύστημα επαγρύπνησης, προειδοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πλέον τα απαραίτητα αυτά σήματα τα οποία θα συνοδεύουν κάποια ιστοσελίδε, σήματα τα οποία ουσιαστικά θα καταδεικνύουν ότι μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αξιόπιστη και το καθεξής. Το ζήτημα πάντω θα πρέπει σίγουρα να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. Περίπου πριν από 100 χρόνια ο Άμπραχαμ Λίνκομ λέγεται ότι το είπε, ορισμένοι λένε ότι το είπε κάποιο άλλο. Αλλά τέλος πάντων, κάποιος είπε πριν από 100 χρόνια ότι μπορείτε να ξεγελάσετε τους πάντες κάποια στιγμή, ορισμένους συνεχώς, αλλά δεν μπορείτε να τους ξεγελάτε όλους και πάντα. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, να έχουμε εμπιστοσύνη στην κοινή λογική. Οι ψευδείς ειδήσει είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αλλά τον έχουμε και ένα Υπουργείο αλήθεια, αν θέλετε, είναι ακόμα χειρότερο. Και πιστέψτε με, εγώ ζούσα σε μια χώρα που είχε τέτοιου είδους Υπουργεία. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, πρέπει να σα πω ότι το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων δεν είναι πρόβλημα μόνο εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μεγάλε αμερικανικέ επιχειρήσει Συγγνώμη, αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στο copyright και στην αμοιβή των καλλιτεχνών. Τέτοια προβλήματα έχουν ε, λοιπόν και στις Ηνωμένε Πολιτείε και εκεί η μουσική λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις αμοιβέ του, ότι είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τα χρήματα τα οποία κερδίζουν μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι τουλάχιστον εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε ακριβώς τέτοια ζητήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίσουν και οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όσον αφορά τώρα το δικαιολογημένο και μη δικαιολογημένο γεωγραφικό αποκλεισμό. όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του τύπου και το καθεξής. Πολλά ζητήματα. Φίξτε, θα συναφερθώ πρώτα στον γεωγραφικό αποκλεισμό. Δεν νομίζω ότι ο αποκλεισμό αυτός είναι δικαιολογημένος όταν ένα 36% όσων θέλουν να αγοράσουν απτά αγαθά από ένα άλλο κράτος μέλος μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αγορά αυτή. Το ποσοστό είναι χαμηλό. Αν εγώ για παράδειγμα θέλω να αγοράσω αυτό το μπουκάλι νερό εδώ πέρα στο Βέλγιο θα πρέπει να μπορώ να εμπιστεύομαι την μάρκα αυτή που μου λέει ότι ε, το νερό αυτό έχει μηδέν θερμίδες. Θα πρέπει να μπορώ και από την Εσθονία να αγοράσω το, το μπουκάλι αυτό νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν, είναι ποτέ δυνατόν όμως να αποδεχθούμε ότι στα πλαίσια τη ενιαία αγοράς ότι κάποιο θα μου πει «Α, όχι, βλέπω ότι εσύ πα να αγοράσει από την Εστονία και δεν σου επιτρέπω να αγοράσει να μπουκάλι νερό από το Βέλγιο». Θα ήταν τεράστιο το σκάνδαλο αν κάποιο δεν μου επέτρεπε εμένα, όντα στην Εστονία, να αγοράσω αυτό το μπουκάλι νερό από το Βέλγιο. Όμω θέλω να αγοράσω αγαθά και υπηρεσίες ε, από κάποια άλλη χώρα, αν τα αγαθά και υπηρεσίες αυτά είναι επιγραμμικά. Και αν κάποιος μου πει όχι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πρέπει να θεωρήσω ότι αυτό είναι δικαιολογημένο. Όχι βέβαια, ούτε και τότε είναι δικαιολογημένο. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θεωρούν ότι υποφελούνται περισσότερο από μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη και όταν θα υπάρχουν διαφορετικές τιμές από περιοχή σε περιοχή, από τη μία χώρα στην άλλη. Όταν εμείς ασχοληθήκαμε με το ζήτημα του γεωγραφικού αποκλεισμού, δεν είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε κοινέ τιμέ παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε ισότιμη μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών όταν θέλουν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίε. Αναφέρουμε αυτή τη στιγμή και στην περίπτωση των παθητικών πωλήσεων αν εγώ για παράδειγμα θέλω να αγοράσω, όπως σας είπα, αυτό το μπουκάλι νερό. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μπορεί να γίνει, γιατί διαφορετικά θα είναι καθαρή διακριτική μεταχείριση. Αν κάποιος μου πει η πιστοτική σου κάρτα είναι στονική και εσύ όντας εστονός ή με στονική πιστοτική κάρτα δεν μπορείς να αγοράσεις αυτό το μπουκάλι νερό. Αυτό το μπουκάλι νερό προορίζεται μόνο για τους δικούς μας τους ανθρώπους, τους δικούς μας τους πολίτες. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της εδαφικότητας, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές και το παραλαμβάνω συνεχώς. Πρέπει να προστατεύσουμε την αρχή της εδαφικότητος. Εγώ έρχομαι από μια μικρή χώρα, την Εσθονία, Και όπως γνωρίζετε, παράγουμε και εμείς ταινίες στη μικρή αυτή την Εσθονία. Και πριν από δύο χρόνια η ταινία Τάντζαριν ήταν υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερη ξένη ταινία. Δεν το πήραμε το Όσκαρ, παρόλα αυτά ήμασταν υποψήφοι, η ταινία είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα υπήρχε κάποιο επιχειρηματικό συμφέρον για κάποιον να αγοράσει τη μικρή αυτή ταινία και την διανύμει σε όλου του κινηματογράφου τη Ευρώπη το επιχειρηματικό συμφέρον ενδεχομένως να εντοπίζεται αν θέλετε στην Εστονία, στις ε, όμορες περιοχές και αξιαγορά περιορίζεται εκεί πέρα. Ενδεχομένως ε, κάποιοι περίεργοι τύποι να θέλουν να δουν την ταινία αυτή από την Εστονία σε μια άλλη, πανευρωπα... σε μια άλλη απομακρυσμένη χώρα και να πρέπει τότε να ε, κάνουν αίτηση για αυτή την πανευρωπαϊκή άδεια, προκειμένου να μπορούν δηλαδή να διανύμουν την ταινία αυτή και σε χώρε εκτό Εστονία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η αρχή τη εδαφικότητα θα πρέπει να παραμείνει, να διατηρηθεί. Σε ένα Δανέζικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου συνάντησα έναν Δανέζο σεναριογράφο και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα, το έχω ξαναπεί αυτό στο παρελθόν. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το Κινηματογραφικό Ινστιτούτο στην Κοπενχάγη και συνάντησα εκεί πέρα Κυρία καθόταν στα δεξιά μου, ένας κύριος καθόταν στα αριστερά μου. Η κυρία αυτή είναι μια πολύ διάσημη σεναριογράφος και έβγαλε έναν καταπληκτικό λόγο. Είπε ότι αγόρασε ένα καταπληκτικό κόκκινο φόρεμα από ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών και το πλήρωσε μόνο 30 ευρώ. 30 μόνο ευρώ το καταπληκτικό αυτοκόκκινο φόρεμα που φορούσε. Είπε ότι το πρώτο της αυτοκίνητο ήταν ένα από τα παλιότερα και πιο άσχημα αυτοκίνητα της Κοπενχάγης. Είπε επίση ε, ότι ε, μολονότι είχε πάρει πάρα πολλά δάνεια, κατάφερε να τα αποπληρώσει πάρα πολύ γρήγορα, το βασικό της μήνυμα πάντως ήταν σαφές. Αλλάξτε το σύστημα. Η συγγραφή είπε δεν λαμβάνουν δίκαια αμοιβή για το έργο τους και όλοι την, την καταχειροκρότησαν. Ο κύριος που καθόταν στα αριστερά μου στη συνέχεια φορούσε ένα κουστούμι το οποίο βέβαια δεν ήταν των 30 ευρώ, ήταν πολύ καλαντημένος και ο τύπος αυτός είπε κάτω τα χέρια από το εφιστάμενο σύστημα βραντικών δικαιωμάτων. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και αυτόν όμω το καταχειροκρότησαν. Και εγώ μετά σκέφτηκα, μα καλά τι κάνω εδώ, γιατί κάθομαι εδώ. Μήπως θα πρέπει οι δύο αυτοί να συζητήσουν πρώτα μεταξύ τους τα ζητήματα αυτά, να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία και μήπως εγώ συζητώντας μαζί τους μετά θα μπορούσα να προτείνω κάτι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πάντως πρόβλημα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όταν μιλάμε για το μη δικαιολογημένο γεωγραφικό αποκλεισμό, ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι υποσχέθηκαν ως επενδυτές απόλυτη γεωγραφική αποκλειστικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι έντιμοι, δεν είναι 100% έντιμοι άνθρωποι. Πω, πώς περνάει ο χρόνος ε, και έχουμε και δεύτερο γύρο ερωτήσεων, έτσι δεν είναι. Το 20% των χρηστών διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν το VPN για να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Το 68% βλέπουν ταινίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχουν πει ότι χρησιμοποιούνται δωρεάν downloads, δηλαδή torrents βασικά, βλέπουν πειρατικά ταινίε. Πολύ, πολύ εύκολα χρησιμοποιεί κανεί το VPN ή το torrent εντελώ δωρεάν. Για του απλού πολίτε δεν είναι πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Είναι μεγάλο πρόβλημα όμω για του δημιουργού, οι οποίοι δεν αμείβονται σωστά βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο. Η απόλυτη λοιπόν εδαφική αποκλειστικότητα, η απόλυτη αποκλειστικότητα ουσιαστικά σε τι αντιστοιχεί, στο 0% ή στο 100%. Αν όμως είναι κάτι μεταξύ των δύο, δηλαδή 20%, 60%, 68%, ε, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για απόλυτη αποκλειστικότητα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πού είμαστε, πώς έχουν τα πράγματα και πού θέλουμε να πάμε. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή με τη δική μας τη στάση να σπρώχνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες προς την πειρατεία. Αντίθετα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές προστατευμένο περιβάλλον για το ψηφιακό αυτό περιβάλλον. Δεν λέει ότι θα πρέπει παντού όλα να είναι δωρεάν και ανοιχτά σε όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομικές αν θέλετε οδούς, μια ε, νομική πρόσβαση προκειμένου να νόμιμη, με συγχωρείτε, πρόσβαση σε ελεύθερο περιεχόμενο. Και αυτό θα πρέπει κάπως να το δούμε, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Έχω μιλήσει για παράδειγμα με ηθήνοντες τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία για τις ταινιοθήκες, τις αρχαιοθήκες, τις οπτικοακουστικές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χιλιάδες ψηφιακά αρχεία και ουσιαστικά υπάρχει και ένα κάποιο ενδιαφέρον από τους πολίτες για τα ψηφιακά αυτά οπτικοακουστικά αρχεία. Υπάρχουν πολλοί πολίτε στι χώρε αυτέ που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και το ίδιο ισχύει εν γέννη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή όμω, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν σε κάποιε χώρε, υπάρχουν πολίτε που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση όπω θα έπρεπε να είχαν σε αυτέ τι ταινίε, σε αυτό το ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει λόγο η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να είναι κλειδωμένη σε αρχεία. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ελεύθερη προ του Ευρωπαίου πολίτε. Αυτό λοιπόν ο στόχο μα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τα φυστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στραφούμε κατά τη αρχή ε, τη εδαφικότητος, θέλουμε να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο για τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ παράλληλα θέλουμε να διασφαλίσουμε και μία δίκαιη κατάλληλη αμοιβή για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Και θεωρώ ότι είναι δυνατό να εξισορροπήσουμε και τις δύο πτυχές. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος έχει πλέον εξαντληθεί, θα επανέλθω στο θέμα της ελευθερίας έκφρασης πριν τελειώσω. Ξέρουμε ότι μετά από κάθε τρομοκρατική επίθεση τα θέματα αυτά επανέρχονται όπως επανέρχεται και η πρόταση να ρυθμίσουμε το διαδίκτυο, να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, παρακολούθησης, έλεγχος. Αλλά βέβαια υπάρχει και η αντίστοιχη πρόταση για προστασία της ελευθερίας έκφρασης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν με εξισορροπημένο τρόπο. Η Γιάννα Τουρμ αναφέρθηκε στην πολυμορφία, στο μεγάλο φάσμα επιλογών που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Όλη η ζωή μας πλέον περνάει από το διαδίκτυο. Είμαστε ψηφιοποιημένοι εντελώς. Και είναι αδύνατον να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, βεβαίως, με τις διάφορες αρμόδιες επιτροπές, με τα κράτη-μέλη και η συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την αρχή της εδαφικότητας, νομίζω ότι απάντησα σε αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την αρχή της εδαφικότητας. Πολιστική πολυμορφία, το έθιξα και αυτό. Πιστεύω ότι το φάσμα των δυνατοτήτων είναι πολύ μεγάλο για να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, το θέμα της, του κυβερνοχώρου, της κυβερνοασφάλειας. Ίσως στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε πρέπει να προβλεφθεί το θέμα αυτό και κάποια άλλα εξάλλου θέματα. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληρέστατες αποφα... Ε, απαντήσεις που μας δώσετε. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερο γύρο γιατί έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας. Ξέρω ότι σας περιμένουν οι υπουργοί από την Ιαπωνία. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να καθυστερήσετε, θα το θεωρήσουν πάρα πολύ προσβλητικό. Πολλά όμως θέματα έχουν μείνει εδώ προς συζήτηση. Ελπίζω πολύ σύντομα να επανέλθετε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας εύχομαι κάθε καλό, καλή επιτυχία στην Προεδρία της χώρας σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Και θα περάσουμε στο επόμενο και το τελευταίο σημείο, όχι μόνο της σημερινής ε, συνεδρίασης, αλλά της τελευταίας συνεδρίασης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε ζητήσει τη μελέτη για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και έχουμε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα αυτής της μελέτης έχει ολοκληρωθεί από τον δόκτορα Μάρκος Προύτς και βεβαίως είναι εδώ με την παλιά του ιδιότητα, ήταν μέλος της γραμματείας μας και φυσικά θα του δώσω τη δυνατότητα να μας κάνει την παρουσίασή του. Το έχουμε το κείμενο του γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Θα ήθελα όμως προηγουμένως να χαιρετήσω τον Ρούπερτ Μέσιος, νέο μέλος της ε, Επιτροπής Πολιτισμού, ουσιαστικά παίρνει τη θέση του Εντολουάν. Μάρκος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ και που δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μου που αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν θα πάω σε λεπτομέρειες επί της μεθοδολογικής προσέγγισης, ούτε θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά που έχω να σας κάνω μια πλήρη σύνοψη. Θα εστιαστώ στα αποτελέσματα της έρευνας και τις συστάσεις που απορρέουν. Απλώς πριν από αυτά θα πω λίγα λόγια για το σκεπτικό, το βασικό άξονα της έρευνας. Υπάρχουν λοιπόν τρία ερωτήματα ερευνητικά που προσπαθώ να απαντήσω στη μελέτη τι είναι η συλλογική ταυτότητα, καταρχάς, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ποιες πολιτικές ακολουθούνται ώστε να ενισχύσουν αυτήν την ευρωπαϊκή αίσθηση της συλλογικής οντότητας. Επίσης, ποιες είναι οι προοπτικές μιας διεθνικής ταυτότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια μη εξελικτική ανάλυση, αυτό το έγγραφο που έχετε μπροστά σας. Προσπάθησα απλώς να κάνω μια συλλογή των επιστημονικών μελετών που έχουν γίνει στο πεδίο αυτό και τις βασικότερες προκλήσεις του σκεπτικού μιας ε, κοινή ευρωπαϊκής ταυτότητας, εστιαζόμενος στον δυνητικό ρόλο της ιστορικής μνήμης, το οποίο με οδηγεί στα βασικά πορίσματα και συστάσεις που συνοψίζονται σε οκτώ σημεία. Πρώτον, η ταυτότητα είναι μια φευγαλία, αλλά αλλά και κονστρουκτιβιστική, λέει ο μιλητής. υπάρχουν πολυεθνικές προσπάθειες τέτοιες όπως είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η ταυτότητα αναλαμβάνει τη σχέση ενός ατόμου με συγκεκριμένες ομάδες ή με το σύνολο της κοινωνίας, επομένως άπτεται των θεμελιωδών θεμάτων του τι είναι το σύνολο της κοινωνίας. Ταυτοχρόνως φαίνεται ότι είναι μια έννοια που οδηγεί σε πολλές διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Εάν υπάρχει κοινό τόπος στην σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση, ακαδημαϊκή προσέγγιση, είναι ότι ταυτότητα δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά δυναμικό και οικοδομημένο. Αυτό ιδιαίτερα για συλλογικές ταυτότητες συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εκείνων οντοτήτων που περισσότερο συνδέονται με μια συλλογική ταυτότητα όπως τα κράτη-έθνη είχαμε και την περίφημη ε, ρίση ενός ερευνητή οι φανταστικές κοινωνίες, οι φανταστικές κοινότητες. Και αυτό εδράζεται στην έννοια της ταυτότητας. Ταυτόχρονα, οι κοινότητες δεν είναι κάτι που φανταζόμαστε μόνο και οι ταυτότητες δεν είναι σταθερές σύν το χρόνο. Και δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα που να είναι ανώτερη μιας άλλης ούτε κάποια ταυτότητα που πρέπει να παραμείνει για πάντοτε. Όμως, η συλλογική ταυτότητα είναι σημαντική. Πάντοτε τη φαντάζεται κανείς, αλλά δεν είναι κάτι το άσχετο. Παρέχει προσανατολισμούς για τους ατόμους, αλλά και για τις πολιτικές κοινότητες, δημιουργώντας αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς μια ομοιότητα που τονίζει ή υποτονίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες των ατόμων σε μια κοινότητα. Κάτι που αν δεν γίνει δεν μπορούμε να μιλούμε για κοινότητα. Σε πολιτικό επίπεδο θα ήταν παράλογο τα κράτη-έθνη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ακολουθούσαν καμία πολιτική ταυτότητας, γιατί τότε δεν θα αναγνώριζαν τον εαυτόν τους ως πολιτική κοινότητα. Σε υπερεθνικό λοιπόν επίπεδο, ποια είναι τα όρια της ανάπτυξης της ταυτότητας. και τι δυνατότητες υπάρχουν. Πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο του ε, κράτους έθνους σε μια δομή σαν εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ γίνεται σαφές ότι ο αντίκτυπος σε υπερεθνικό επίπεδο μια έννοια όπως είναι η ταυτότητα έχει και δυνατότητε και κινδύνους. Το κράτος έθνος είναι ένα βασικό σημείο αναφοράς για την έννοια της υπερεθνικής ταυτότητας. Τα ισχυρά έθνη είναι οπωσδήποτε ένας παράγοντας που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τους και παράλληλα είναι και ένα από τα λίγα διαθέσιμα μοντέλα, πρότυπα, για τον συνδυασμό ετερογενών κοινωνικών ομάδων σε μία κοινότητα. Ο κίνδυνος είναι ότι γίνονται συγκρίσεις ή αναλογίες εκεί όπου καμιά φορά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό γιατί η αντίστοιχη έννοια σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμη. Επομένως, οι εθνικές ταυτότητες δεν μπορούν να είναι το απόλυτο πρότυπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι τα εθνικά πρότυπα δεν έχουν καμία χρήση, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα προς ένα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Επομένως, ποια θα μπορούσε να είναι η ουσία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Εδώ θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι μια τέτοια ταυτότητα πρέπει να είναι και πολιτική και πολιτιστική. Στην Ακαδημία συχνά κάνουμε μία διάκριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινή κοινότητα αξιών ή κοινή κοινότητα δημοκρατικών πρακτικών το οποίο για τους γερμανόφωνους ε, συνδυάζεται με κάποιες έννοιες που είχε αναπτύξει ο Χάμπερμας και τις πολιτιστικές ταυτότητες στις οποίες αναφερόταν. Πολύ συχνά η ταυτότητα θα μπορούσε να είναι άθροισμα των εθνικών προτύπων με όλα τους τα προβλήματα. Πρέπει να ορίσει κανείς τι είναι αυτό που τον κάνει να ανήκει σε μια κοινότητα. Αλλά έχουμε και εμπειρικά ερωτήματα τι κάνει κανείς με την διαφορετικότητα αν θέλει κανείς να αναπτύξει πολιτιστική ταυτότητα. Και η πολιτική κοινότητα βεβαίω έχει περιορισμούς. Πολλοί την βλέπουν ως μια έννοια ελιτιστική και αφηρημένη ή τη βλέπουν ακόμα και ως πολιτική ζήλου, το οποίο καμιά φορά ταυτίζεται με τα εθνικά πρότυπα ταυτότητας. Τι είναι λοιπόν κάτι, τι είναι αυτό που σε κάνει να ανήκει σε μια κοινότητα και να μην ανήκει σε μια άλλη κοινότητα, το οποίο ισχύει και για θρησκευτικές ομάδες. Επομένως χρειαζόμαστε μια ταυτότητα που να είναι ορίσιμη πολιτιστικά, αλλά και να οδηγεί σε μια δημοκρατική κοινότητα εστιασμένη στους πολίτες. Σε ποιο βαθμό λοιπόν οι πολιτικές της Ένωσης μας βοηθούν για μια τέτοια κοινή κατανόηση. Αυτό που εδώ πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω. Οι πολιτικές ταυτότητες ακολουθούνται από την αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά ασυνεπώς και κατακυρισματισμένα και με διαφορετική ένταση στα χρόνια. Αυτό είχε να κάνει με διάφορες επικρίσεις που υποβάλλονταν, αλλά και από την εντύπωση ότι οι πολιτικές ταυτότητες ήταν από πάνω προς τα κάτω εφαρμοσμένες. Υπό την έννοια αυτή, το πρόγραμμα Europe for Citizens προσπαθεί να υλοποιήσει μια αλλαγή παραδείγματος, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Όπως βέβαια γνωρίζουμε όλοι, δεδομένων των χρηματοδοτικών και άλλων περιορισμών, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αντίκτυπο επί του συνόλου των πολιτών, αν θέλουμε να αναδειχθεί κάτι σαν ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από τις πολιτικές. Και αυτό είναι σημαντικό και σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών ομελών ακόμα περισσότερο αν επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο ποδίο, πεδίο πολιτικής, η ιστορία ίσως είναι τέτοιο επίπεδο που ήταν πεδίο αντιπαραθέσεων στο παρελθόν αλλά και δυνητικής συνένωσης για το μέλλον. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως επί του παρελθόντος είναι δύσκολο να ζούμε στο παρόν και πολύ ακόμα περισσότερο δύσκολο να φανταστούμε το κοινό μέλλον. Αυτή λοιπόν η ποικιλομορφία, η διαφορετικότητα των ιστορικών παρελθόντων είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ίσως να μην συμφωνούμε όλοι σε μια κοινή ερμηνεία των ιστοριών ή της ιστορίας ή του παρελθόντος, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Δηλαδή, αντί να μην μιλούμε αντί να μιλούμε μάλλον για μια πολιτική μνήμης ιστορικής, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια προσέγγιση του πώς σκεπτόμαστε το παρελθόν από κοινού, του πώς αποτυπώνεται αυτό στις βασικές αρχές των συνθήκων και χωρίς αυτό να βασίζεται σε μια προκατασκευασμένη εικόνα ερμηνεία του παρελθόντος, αλλά ενός ανοιχτού βήματος διαλόγου αναγνωρίζοντας τα ιστορικά γεγονότα ως στοιχεία αξιολόγησης και απομακρυνόμενοι από την έννοια ότι υπάρχει μία ιστορική πραγματικότητα, μία ιστορική αλήθεια. Υπάρχουν διάφορα ιστορικά γεγονότα, αλλά δεν υπάρχει ενιαία πραγματικότητα που να μπορεί να ισχύει για όλους. Επομένως, μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει μια κοινή αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα, το οποίο με οδηγεί στο τελευταίο από τα σημεία των πορισμάτων. Προκειμένου να πετύχουμε κάτι τέτοιο, ο ρόλος της παιδείας είναι θεμελιώδης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα σε επίπεδο σχολικής παιδείας είναι να εξασφαλίσουμε ποιοτική διδαχή της ιστορίας και να δώσουμε τα μέσα στους διδάσκοντες να αναλύουν και να εξετάζουν τα γεγονότα του παρελθόντος σε ένα ευρύτερο πεδίο. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να είναι πιο επικριτικοί στην εθνική τους, αν θέλετε, η προσωπική τους ιστορία. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατάρτιση και εκπαίδευση και των διδασκάλων. Το οποίο, προφανώς πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο προσέγγισης για την εκπαίδευση. Χρειάζεται αντίστοιχα λοιπόν να έχει κανείς υλοποιήσει τα διάφορα επίπεδα της πολιτικής παιδείας του. Όπως και μια, έναν πολιτισμό, αν θέλετε, του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών μέσω της προαγωγής προγραμμάτων όπως το Εράσμους προκειμένου να γνωρίσει κανείς τη διαφορετικότητα την πολιτιστική που υπάρχει στην Ευρώπη. Να τολμάει κανείς δηλαδή να γνωρίσει προκειμένου να συμπεράνει. Το οποίο με οδηγεί σε κάποια σε κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Καταρχάς χρειαζόμαστε ένα κοινό με κριτική ικανότητα, με συμμετοχή των πολιτών σε μια κοινή ευθύνη για το βασικό άξονα της πολιτικής, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό πεδίο, ώστε να ανακύψει μια τέτοια κοινότητα πολιτών. Κατά πόσον μια ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών θα δώσει τελικά μια κατεύθυνση ευρωπαϊκής ταυτότητας, μένει να το δούμε. Πέραν του ερωτήματος τι είναι η Ευρώπη και πού πηγαίνει, που ίσως είναι αρκετά επίγον σήμερα, δεν φαίνεται να είναι φτωχή η συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας σήμερα. Δεν έχουμε μία ενιαία γλώσσα ή ενιαίο πολιτισμό. και δεν μπορούν δηλαδή υπό την έννοια αυτή να μεταλαμπαδευτούν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χρειάζεται ένα συνδετικός κρίκος το οποίο μας οδηγεί σε ένα παράδοξο. Ένα από τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η επιφυλακτική και προσεκτική στάση που διατηρεί απέναντι στον Ιμπεριαλισμό που κυριαρχούσε στην ευρωπαϊκή σκηνή στο 10ο αιώνα, 9ο και αρχές του 20ου αιώνα. Στην απομάκρυνση από τις σαφείς διακρίσεις φίλοι-εχθροί. το παράδοξο είναι ότι αυτό την ίδια στιγμή είναι και ο μεγαλύτερος περιορισμός της. Είναι όμως κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Δεν υπάρχει σαφή απάντηση σε αυτό. Δεν είναι στόχος ε, καθεαυτός η επίτευξη ή η κοινή αναγνώριση μια τέτοια ταυτότητα, όλα εξαρτώνται από το είδος της κοινότητας ή της κοινωνίας που θα θεωρήσουμε πιο επιθυμητό σε κάθε χρονική στιγμή. Χρειάζεται ένα, ένα σύστημα αξιών, μια οικογένεια, μια τοπική κοινότητα, ένα έθνος ή μια ευρωπαϊκή κοινότητα που να συνενώνει και όχι να διαιρεί. Αλλά το τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει σχετικά με την ε, αντίληψη που έχει κανείς σχετικά με την ταυτότητα. Έχουμε ήδη πολλαπλές ταυτότητες που ισχύουν, που υφίστανται παράλληλα σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, χωρίς η μία να μειώνει την άλλη. Δεν υπάρχει λοιπόν πιστικό επιχείρημα γιατί η σημερινή πολλαπλότητα ταυτοτήτων δεν θα μπορούσε να συμπληρωθεί ή να εμπλουτιστεί με ένα πρόσθετο επίπεδο ταυτοποίησης, είτε το ονομάσουμε ευρωπαϊκό είτε κοσμοπολιτικό. Αν θα μπορούσαμε να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα όχι ως κάτι που κινδυνεύουμε να χάσουμε, αλλά κάτι που ίσως να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για σχεδόν φιλοσοφική συζήτηση. Είναι εξαιρετικό το θέμα, το θέμα της ταυτότητας δεν μπορεί να επιβληθεί εκ των άνω, πρέπει σιγά σιγά να δημιουργηθεί, να προκύψει και αυτό που είπατε στο τέλος είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει κάποιος να είναι ευτυχής αν έχει πολλές ταυτότητες. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, είναι αυτό που με ορίζει σε σχέση με τους άλλους που με ξεχωρίζει. Μπορεί κάποιος να είναι ριζωμένος σε μια περιοχή, να ανήκει σε αυτή, να έχει όμως και μια ταυτότητα περιφερειακή, τοπική, ε, εθνική, αλλά να είναι και Ευρωπαίος. Όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά. Και συνήθως θεωρούμε ότι η ταυτότητα είναι κάτι που αφορά την πατρίδα. Στη Γερμανία δηλαδή πολλές φορές ε, το ταυτίζουμε. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, είναι αυτό που μας ε, κάνει να νιώθουμε άνετα στο σπίτι μας. Αλλά μπορεί κάποιος και σε μια μικρή μονάδα να νιώσει άνετα στην οικογένειά του παραδείγματο χάρη. Ή μπορεί εγώ να νιώσω ότι είμαι άνετα και νιώθω σπίτι μου και στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά. Είναι κάτι το οποίο και εσείς αναφέρατε. Ότι δηλαδή το ότι ταυτιζόμαστε με τη δημοκρατία, με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις δημοκρατικές αξίες, αυτό είναι κάτι που συναποτελεί την ταυτότητά μας και είναι συνιστόσα της ταυτότητάς μας. Είναι κάτι που δεν μπορεί αυτόματα, δηλαδή, να σημαίνει εθνικό χαρακτηριστικό. Πώς μπορεί κάποιος να ταυτοποιηθεί με δημοκρατικές αξίες, να συνειδητοποιήσει ότι ανήκει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι μια κοινότητα που σέβεται και δέχεται τις δημοκρατικές διαδικασίες και όχι την πατρίδα που πολλές φορές μπορεί να ταυτιστεί και με κάτι διαφορετικό, με το στρατό, η εκπαίδευση επίσης είναι ένα χαρακτηριστικό με το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε την ταυτότητά μας. Σε κάθε περίπτωση όμως η ταυτότητα δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας ορίζει και μας ξεχωρίζει από τους άλλους. Μπορεί να είναι και κάτι που έχουμε κοινό με τους άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μελέτη κοιτάω γιατί πιστεύω ότι αυτή η μελέτη μπορεί καθημερινά να μας εμπνεύσει. Νομίζω ότι το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι κάτι που πρέπει να το επεξεργαστούμε, κάτι που ενδεχομένως θέλουμε να το ορίσουμε καλύτερα και για το οποίο θέλουμε να πολεμήσουμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η μελέτη σας. Μας δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι μια έννοια που δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάθος και με υπερβολική φόρτιση. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ζω σε μια χώρα που σύντομα θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο χρόνια συγκεκριμένα. Επομένως υπάρχουν αυτές οι επικαλυπτόμενες ταυτότητες στις οποίες αναφερθήκατε με Άγγλος, Βρετανός και Ευρωπαίος. Και ε, ανήκω στην Ευρωπαϊκή Διασπορά επίσης. Υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων, αν θέλετε, οι αρχές, οι απαρχές βρίσκονται στην Ευρώπη, αναφέρομαι στον Καναδά ή σε άλλες χώρες. Επομένως, το ερώτημά μου το ακόλουθο. Σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή ταυτότητα που αισθάνεται ένα άτομο εξαρτάται τελικά από τον τόπο που διαμένουν, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για χώρε Ευρώπη που βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ή για χώρε οι οποίε είναι εκτό Ευρώπη αλλά οι οποίε είναι πάρα πολύ συγγενικέ με την Ευρώπη, έχουν προέλθει από την Ευρώπη αν θέλετε. Ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Μάλινοφ, αν ήταν ακαδημαϊκή θεωρητική συζήτηση και αν βρισκόμασταν τώρα σαν ένα πανεπιστήμιο και αν συζητούσαμε μία διατριβή διοκτορά, τότε προφανώς εγώ θα έλεγα στην Κρητική Επιτροπή σίγουρα να δώσει τελικά το δακτορικό με τον καλύτερο δυνατό βαθμό στον ε, συντάκτη της έκθεσης αυτής, της μελέτης, της διατριβής αν θέλετε, γιατί ε, είδαμε αυτή τη στιγμή ότι αναφέρατε πάρα πάρα πολλούς ε, σημαντικούς στοχαστές, Χάμπερμας και πολλούς άλλους. Πάντως, πρέπει να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μου έκανε εντύπωση ότι το νέο μέλος της Επιτροπής έθεσε το ερώτημα το οποίο ήθελα να θέσω εγώ από πολιτικής πλευράς. Αν εγώ συμμετέχω σε μια πολιτική συζήτηση, πώς θα πρέπει να απαντήσω σε κάποιον ο οποίος μου λέει αγαπώ την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα πολιτικής φύσης αν θέλετε που έχω και που θα ήθελα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος είναι ο γενικότερος πολιτικός στόχος της μελέτης σας, ποια είναι η πολιτική προσέγγισή σας, το να καταφέρουμε να προασπίσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι να προασπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτός είναι ο απότερος στόχος της μελέτης σας, τότε θα ήθελα να γνωρίζω τι έμπρακτα μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική και εδώ πέρα σχεδόν αναφέρομαι σε αυτό που είπατε για τον Αβραάμ Λίνκολ. Διαφορετικά μπορούμε να μιλάμε συνεχώς για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και αυτό το επιχείρημα, εφόσον υποθεί, θα είναι και πάρα πολύ ισχυρό. Αλλά δεν θέλουμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αν να προσπίσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυτός είναι ο πολιτικός σας στόχος, τότε διαφορετική θα πρέπει να είναι η προσέγγιση και συγχαρητήρια γιατί καταφέρετε να ξεπεράσατε ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Το να εγκαταλείψουμε το νεολογικό πλαίσιο το, του έθνου κράτους κάθε φορά που μιλάμε για την ταυτότητα, τη δημοκρατία και το καθεξής. Πάντως νομίζω ότι η βάση της μελέτης σας είναι πολύ καλή. Και ίσως αυτό που είπατε, overcoming history, να καταφέρουμε να υπερβούμε τελικά την ιστορία, ίσως αυτό να είναι το πιο κεντρικό στοιχείο. Το να υπερβούμε την ιστορία δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την ιστορία, ότι διαφορούμε για την ιστορία. Σημαίνει ότι κάνουμε μια συνειδητή διανοητική προσπάθεια. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα όταν διάβαζα τη μελέτη σας. Πώς θα καταφέρουμε να υπερβούμε την ιστορία. Overcoming history. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Επομένω, δεν είναι σχεδόν φιλοσοφική συζήτηση, είναι σαφώ φιλοσοφική συζήτηση. Είναι η πιο φιλοσοφική συζήτηση που έχω κάνει ποτέ στην Επιτροπή αυτή. Äh, ναι. Όντω, έτσι είναι μάλλον. Μάρκου. Να προσθέσω κι εγώ τις δικές μου ευχαριστίες και εκτίμηση για αυτήν την πληρέστατη και πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και αναφέραμε και στη βιβλιογραφία που έχετε προσθέσει εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η διάκριση στην ερώτηση της ταυτότητας μεταξύ μιας πολιτιστικής ταυτότητας κοινών αξιών και μιας πολιτικής κοινότητος που είναι επίσης επί τη βάση βεβαίως και πάλι κοινών δημοκρατικών αξιών. Μου φαίνεται μια διάκριση πάρα πολύ χρήσιμοι ώστε να αναπτυχθούν ε, εκ παραλίλου τις ε, προσεγγίσεις που πρέπει ε, να έχουμε προκειμένου να κάνουμε την τελική σύνθεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων ώστε να φτάσουμε σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ήθελα και εγώ απλώς να σημειώσω δύο στοιχεία που θα, ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Θεωρώ ότι ο πυρήνας των αξιών δεν είναι μόνο αυτός που αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν ή στην ιστορία, αλλά είναι κάτι στο οποίο έχουμε φτάσει και ίσως δεχόμαστε από κοινού όπως λέτε μετά από πάρα πολλές μετεξελίξεις φιλοσοφικές, ιστορικές και θεωρητικές. Αυτός ο πυρήνας αξιών λοιπόν δεν θα έπρεπε να τοποθετείται κατά την άποψή μου μόνο στο πεδίο της μνήμης, αλλά σε ένα πεδίο συνεχούς εκπαίδευσης. Όπως λέτε πολύ ωραία για τις υπόλοιπες έννοιες και οντότητε που είναι δυναμικές και όχι σταθερές, γιατί μια άλλη σημαντική έννοια είναι η συνύπαρξη. Πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε επί τη βάση αυτών των ε, ερμηνεών, αξιών και ενιών. Επίσης μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που συστήνεται σχετικά με τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για να κλείσω. Εσείς τι θεωρείτε ότι ποια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η αποστολή αυτού του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ας πούμε. Τι είδους, πώς θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε τη δουλειά αυτή και όχι μόνο σε σχολικό επίπεδο εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκος, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να απαντήσω. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ερώτησή σας που αφορά την ταυτότητα. Βεβαίως και παίζει ένα καθοριστικό ρόλο το θέμα της περιστασιακής δηλαδή ταυτότητας από πού προέρχεται κάπως αλλά και πού μένει τη συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή που βρίσκεται. Μπορεί κάποιος δηλαδή μπορεί να πάει στην Σκοτία να νιώθει ακόμα πιο Άγγλος ή αν πάτε στη Γαλλία θα νιώσετε ακόμα πιο Βρετανός. Είναι σαφές ότι αλλάζει η ταυτότητα ανάλογα με το με ποιον τρόπο τη βλέπουμε, πώς την αντιλαμβανόμαστε και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η αντίληψη του ευρωπαϊκού χαρακτήρα της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, τι είναι ευρωπαϊκό, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πού μένει κανείς, πού βρίσκεται κανείς. Κύριε Μάλινο, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που με ακούσατε ότι από ακαδημαϊκής απόψεως σας άρεσε η παρουσίασή μου. Όσον αφορά το σκοπό αυτού του κειμένου, εγώ θα σας απογοητεύσω γιατί είχα μια πάρα πολύ μετριοπαθή, ε, ένα πολύ μετριοπαθή στόχο. Ήθελα να καταλάβω αυτό που σχολίασε και η Πρόεδρος, ότι δεν είναι κάτι το αποκλειστικό. ήθελα να αποδείξω ότι δεν είναι κάτι το αρνητικό από μόνο του. Και δεν είναι ο σκοπός μου να προσπιστώ την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δουλειά των πολιτικών. Εγώ ήθελα απλώς να προετοιμάσω το έδαφος για μια ανδεχόμενη συζήτηση. Να δώσω κάποιες φιλοσοφικές έννοιες και να δω ποια είναι τα εμπόδια που προκύπτουν. Την ίδια ώρα, διαβάζοντας το κείμενο, προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δημιουργεί κάποια τέτοια προβλήματα. Ε, το πρόγραμμα Εράσμους, παραδείγματος χάρη, συνεισφέρει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και ακόμα και αν δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το κείμενο. Παρόλα αυτά δίνω κάποια στοιχεία που να ενισχύουν την ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Άρα, ενώ δεν ήταν αρχικά ο σκοπός μου να βρω επιχειρήματα για να προσπιστούμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, ίσως ενδεχομένως κάτι τέτοιο να γίνεται. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε αυτό που είπατε στο τέλος, τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ναι, υπάρχουν συνάδελφοι που προσπάθησαν να το δημιουργήσουν. Ε, η Επιτροπή μας ήταν πραγματικά από αυτούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και αυτό που έγινε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όλη η ευρωπαϊκή ιστορία βρίσκεται σε ένα κτίριο και βεβαίως ενώ υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά είναι πολύ σημαντικό το έργο που έχει γίνει σαν ιστορικός, σαν ε, ειδικό για θέματα πολιτικής και ιστορίας. Θεωρώ ότι υπάρχουν εδώ κάποιες ε, ελλείψεις και αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη είναι η ιστορία των απικιών, οι αυτοκρατορίες, ο εμπεριαλισμός δεν παρουσιάζονται ίσως όπως θα έπρεπε. Αλλά Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα από διαφορετική άποψη και να τα ερμηνεύσουμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους όσους είναι εδώ. Θα τους ε, προτείνουμε το κείμενο της μελέτης σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι και στην πράξη εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού θα μπορέσετε να μας τροφοδοτήσετε με κάποια φιλοσοφικά κίνητρα και κάποια από τα αποτελέσματα των εργασιών σας. Δεν θέλω να ολοκληρώσω τη συνεδρίαση πριν σας πω ότι στις 4 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουμε εκ νέου 3 με 6.30. Σας εύχομαι όλους ένα ονειρεμένο καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε λίγο να ξεκουραστείτε και να μας ξαναέρθετε εδώ με ανανεωμένες δυνάμεις και ενθουσιασμό. Στις 5.30 ε, θα συνεδριάσουν εδώ οι συντονιστές. και ελπίζω να ενημερώσετε τους συντονιστές σας και να είστε ακριβείς. Ακριβώς στις 5.30 θα αρχίσουμε. Έχουμε λίγη δουλίτσα για τους συντονιστές, αλλά όσον αφορά την τακτική συνεδρίαση, ξεκινάνε οι διακοπές μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλές διακοπές.